buenos días. Vamos un poco retrasados. Καλημέρα σα, Έχουμε μια, κάποια καθυστέρηση. Με συγχωρείτε που αργήσαμε, αλλά θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Ανακοινώσεις. Μια πολύ σύντομη. Όπως βλέπετε, έχει υπάρξει μια αλλαγή στην Προεδρία μας. Εδώ δεξιά μου έχω τον νέο τμήματάρχη, κύριο Μάικλ Τόπινγκ ο οποίο ε, ήδη έχει αναλάβει τα καθηκοντά του. καλώ ήρθατε, το είπα και στους συντονιστέ. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία, λοιπόν, πολλή προσπάθεια και πολλή εργασία στις συνεδριάσεις μα. Πρέπει οπωσδήποτε, επειδή έχουμε εδώ τον κύριο Τόπινγκ, σημαίνει ότι κάποιο δεν είναι. Είναι η Μαρίλια Κρέσπο, που όπως είπα προηγουμένω, ήταν τμήματάρχη, επανήλθε, έφυγε και τώρα ενώ επανήλθε ξαναφεύγει. Θέλω να την ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την εργασία την οποία επετέλεσε από τότε που είμαι πρόεδρος της Επιτροπής σας. Εύχομαι κάθε τύχη στις νέες εργασίες, στις οποίες επανέρχεται. Και όπως είπα, όπως πηγαίνω έρχεται, το μόνο που ελπίζω είναι ότι αν θελήσει να επανέλθει, να κάτσει λίγο περισσότερο, διότι η δουλειά μας είναι πολύ δύσκολη, είναι πολύ δουλειά. Ευχαριστούμε τη Μαρίλια και καλώς ήρθες Μάικλ. Έχουμε μια μεγάλη ε, ημερήσια διάταξη ψηφοφοριών, οπότε το πρώτο που ζητάω παρακαλώ είναι λίγη ησυχία. Δεύτερο, παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί, να προσπαθήσω να τις κάνω δηλαδή με το χέρι, για να πάμε πιο γρήγορα. Εντάξει, θα, τις, την κάνουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία ορισμένες φορές. Επειδή όμως, ε, επειδή έχουμε πάρα πολλές ψηφοφορίες, παρακαλώ να πάνετε γρήγορα. Ο κύριος Ασένης, για την ημερήσια διάταξη της Επιτροπής μας, ως εισηγητής για την ομοθεσία για την ε, βαθιά θάλασσα θα ήθελα να αναβάλουμε τη συζήτηση, την παρουσίαση της Επιτροπής για άλλη μια εβδομάδα γιατί μόλις ανέλαβα το θέμα αυτό θα ήθελα να έχω χρόνο να το εξετάσω πριν από την αρχική συζήτηση απέστειλα το αίτημα και γραπτός. Κύριε Στεβέ, κοιτάξτε, ε, θα έπρεπε να καταλάβει ότι πρέπει να συζητηθεί αμέσω το θέμα του κύριου Αρσένη. Α, καλά, για άλλη μια εβδομάδα, εντάξει. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη, εγώ έφτασα. Είναι δικό μου το λάθος. Ε, ε πρέπει να δούμε την έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Έχει δίκιο, είναι το σημείο 14 προτείνει να το αφήσουμε για την επόμενη συνεδρίαση. Ωραία. Μου το είπε, μου το είπε, αλλά άρχισα να μιλάω για και το ξέχασα. Το 14 λοιπόν αναβάλλεται. Το 14. Εντάξει, όπως είπε και η κυρία ε, Φράγα, όπως είπα και απαντώντας στην κυρία Φράγα, οι ψηφοφορίες θα γίνουν όλες η μία μετά την άλλη. Εντάξει, να είναι σαφές αυτό. Γι' αυτό σας το λέω. Θα γίνουν όλοι η μία μετά την άλλη. Όλες τη, η μία μετά την άλλη. Το πρώτο θέμα είναι η έκθεση Λεύιν. για την εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Εντάξει. Έχετε όλοι λοιπόν την... Λοιπόν, έχουμε συμβαστική ένα. Άρχεται λίγη. Είναι ηλεκτρονική. Εγκρίνεται. Τροπολογία 46. Άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. 44. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 45. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 47 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3 άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55. Παρακαλώ, πέστε μου. Υπάρχει μία τροπολογία η οποία έχει διαγραφεί ε, εκεί που λέγεται ε, αυξήσει τον τιμών θα θέλαμε να υπάρχει διακύμανση των τιμών. Ποιο πρόβλημα υπάρχει, λέει ο Πρόεδρος. Ποιο είναι το θέμα, δεν κατάλαβα. Υπάρχει μια τραπολογία του κυρίου Στίβενσον, η 55. Αυτήν ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. είναι το θέμα ότι έχει αλλάξει η διατύπωση στο εσωτερικό της τροπολογίας. Η διατύπωση στο εσωτερικό της τροπολογίας. Α, μάλιστα. Πρόκειται για προφορική τροπολογία λοιπόν, όπου προτείνεται να αλλάξει, αντί να βάλουμε αύξηση της τιμής, να βάλουμε διακύμανση της τιμής. Είναι κανείς που διαφωνεί με αυτήν την αλλαγή. Κανείς. Ωραία. Οπότε είναι ναι, διατυπωμένη διαφορετικά η τροπολογία. Ψηφίζουμε λοιπόν το 55 με την προφορική, με την προφορική της τροπολόγηση. Άρχεται. Πέρασε. Άρχεται λέει ο πρόεδρος. Όχι, λίγη. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τα μηχανήματα γιατί βλέπω μόνο 6. Ξαναρχίζει η ψηφοφορία της τροπολογίας 55. Άρχεται. Λίγοι. Εγκρίνεται. 58 άρχεται. Λίγοι. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 και 4α. Α, πρώτα την 4. Λοιπόν, άρχεται για την 4. Συμβαστική. Λίγη. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Λίγη. Τι υπήρξε πρόβλημα. Α, καλά, όχι, εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Ε, ε, λίγη, συγγνώμη. Εγκρίνεται. 78. Την οποία θα ψηφίσουμε σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Λίγη. εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, ε, άρχεται. Λίγη. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 84. Υπέρ. Ε, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Α, δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Αλλά έχουν ψηφίσει 23 ούτως ή άλλως. Πιανού το μηχάνημα δεν ε, δουλεύει. Εντάξει, δεν, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται ούτως ή άλλως. Συμβαστική 9 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 89 άρχεται πέρας εγκρίνεται 90 άρχεται πέρας εγκρίνεται 91 άρχεται πέρας εγκρίνεται 92 άρχεται πέρας απορρίπτεται Τροπολογία 93. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία είναι τα 10. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία 95. Άρχεται. Πέρας. Τι έγινε. Τροπολογία 95. Άρχεται. Πέρας. Λοιπόν, ξαναρχίζουμε. Άρχεται. 95. Πέρας. Εγκρίνεται. Αχ, πρώτη συνεδρία του με μετά. 96. Άρχεται. πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 104 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 105. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 107 με την ε, προφορική τροπολόγηση. Άρχεται. Όχι, όχι, Ωραία, ψηφίζουμε την 107. Άρχεται. Άρχεται λέω. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, η τροπολογία 107. Άρχεται. Τώρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 106. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 110. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 111. Άρχεται πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 13. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε Καλά δεν παίζει ρόλο στο αποτέλεσμα. 119. 119 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 122 άρχεται. Πέρας. 122. Εγκρίνεται. 124 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. 123. 123 άρχεται. Πέρασε, εγκρίνεται. 125. Άρχεται. 125. Πέρας. Εγκρίνεται. 126-127 ταυτόσημες. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14. Άρχεται. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Έχει δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 134. Άρχεται. 134. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 139. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύε 8. Άρχεται. Α, καταπίπτει βεβαίω. Είναι τα 5. Άρχεται. Είναι τα 5. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 16 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 143 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 15. ΔΕΒΕ 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Άρχεται. Α, δύο τμήματα, δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Και το δεύτερο, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται και αυτό. 149 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 152 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική 18α, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 158 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒ 7. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 19 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 161 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 166 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ντεβε 9 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 168 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 167 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαστική 21 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Σημαστική 22 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 178 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 179 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 183 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 24 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 187 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 188 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 186 άρχεται. πέρα Απορρίπτεται. 190 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 191 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 192 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 14 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 27 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 200 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 28 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 206 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 30 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 215 και 216 ταυτόσημες άρχονται. Πέρας. Απορρίπτονται. Τροπολογία, συγγνώμη, συμβασμός 31. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 221. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 32. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 225. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 226. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 227. Όχι, 228. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε. Το δεύτερο τμήμα αποσύρθηκε έτσι. Θα ψηφίσουμε. Είναι ταυτόσιμη. Ωραία. Αποσύρθηκε λέγεται στον πρόεδρο. Πάμε στην 237 λοιπόν. Ψηφίζουμε την 237. Α, το δεύτερο τμήμα λέτε εσείς. 237 δεύτερο τμήμα. Εντάξει, ψηφίζουμε λοιπόν. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε τώρα την 231. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 230. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 232. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 233. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 235. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 236. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 234. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 238. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 239. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. 240 και 241 είναι ταυτόσιμες από κοινού. Άρχεται, πέρας, απορρίφθηκαν. Συμβιβασμοί 35 και 37. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκαν. Συμβιβασμός 36. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε τροπολογία 247 άρχεται πέρας εγκρίθηκε πάμε στην 240, 255 255 άρχεται πέρας Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. 255 είπαμε. Εγκρίθηκε. 256 τώρα. Άρχεται. Συγγνώμη. Από η 257 τώρα. 257. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 258. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 259 και 260 ταυτόσημες άρχεται πέρας εγκρίθηκαν 264 264 λοιπόν άρχεται πέρας απορρίφθηκε απορρίφθηκε 265 τροπολογία άρχεται πέρας εγκρίθηκε 267 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 268 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 269 άρχεται πέρας επαναλαμβάνουμε 266 διορθώνει ο πρόεδρος. 266 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η 266. Από την ίντα η 6 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. 229 τροπολογία άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. 269 τώρα. 269 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 270 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 271 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 273 άρχεται. Πέρα, ε, πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 274 άρχεται πέρας εγκρίθηκε. 272 άρχεται πέρας εγκρίθηκε. 275 άρχεται πέρας εγκρίθηκε. 276 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 278 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 279 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 280 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 281 άρχεται Πέρας. Εγκρίθηκε. Ίντα εννέα Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ίντα οκτώ Δεύτερο τμήμα. Ίντα οκτώ Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. 282. Άρχεται. Πέρας απορρίφθηκε 283 άρχεται πέρας εγκρίθηκε 284 άρχεται πέρας εγκρίθηκε τροπολογία 1 άρχεται πέρας εγκρίθηκε Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβασμός αιτιολογικής σκέψης α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 9. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 8. Άρχεται. Όχι. Μια και εγκρίθηκε η άλλη. Η 10. Άρχεται. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Καταψηφίστηκε. Συμβιβασμός στην αιτιολογική σκέψη Β. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 18. Άρχεται. Πέρας. Καταψηφίστηκε. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός στην σκέψη Δέλτα. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Συμβιβασμός ε και εα σε ξεχωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε το πρώτο. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε και το δεύτερο τμήμα. Τροπολο... Συμβιβασμός στο σίγμα τάφ, F, άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 35 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα, άρχεται. Πέρας απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 33. Μόνο ένα τμήμα, έτσι. Το πρώτο αποσύρθηκε. Δεύτερο τμήμα της 33. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 36. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 37. Συγγνώμη, 38. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 32. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Εντάξει. Τώρα θα ψηφίσουμε το ψήφισμα όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίθηκε. 24 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια κυρία Λεβίν. Και περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία. Πού είναι... η ψήφιση της μικρής κλίμακας και χειρονακτικής παράκτειας αλίας του κυρίου Φερέιρα έκθεση, σχέδιο έκθεσης. Αν συμφωνείτε ξεκινούμε και συνεχίζουμε ήδη. Hemos cambiado los papeles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 No, no, no, ver, Συγγνώμη, καταπίπτει αφού εγκρίθηκε η προηγούμενη 58. Έτσι καταπίπτει λοιπόν. Η τροπολογία 80 τώρα επειδή καλύφθηκαν οι προηγούμενες. Η τροπολογία 80 τώρα. 80 λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Η 63 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 64 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Περνάμε στον συμβιβασμό 11 λοιπόν, πρώτο τμήμα. Α, εγκρίθη, επειδή εγκρίθηκε η 68 λέτε. Ναι, καταπίπτει, καταπίπτει. Πάμε στην 83, 83 τροπολογία τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία ταυτής. αυτής. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τοπολογία 81. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 13. Πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίφθηκε. Συμβασμός 13 δεύτερο τμήμα άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 78. 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. απορρίφθηκε. Τροπολογία 79. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η 84. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 14. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε η τροπολογία, ο συμβασμός 15 τώρα, άρχεται. Πέρας, εγκρίθηκε. Η τροπολογία 96 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η ισοψηφία απορρίφθηκε. Η τροπολογία 99 άρχεται. Ψηφοφορία. Πέρας απορρίφθηκε. Συμβασμός 16. Πρώτο τμήμα άρχεται. Μάλιστα, πρώτο τμήμα άρχεται, εγκρίθηκε. Συμβασ... Ε, συμβασμός 16, δεύτερο τμήμα άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 97. Η τροπολογία 100. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 100. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 106. Άρχεται. Πέρας απορρίφθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 17. 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 109. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η 110. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 112 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 113 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 114 άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Συμβασμός 18, πρώτο τμήμα, άρχεται. Πέρας, εγκρίθηκε. Συμβασμός 18, δεύτερο τμήμα, άρχεται. Πέρας, εγκρίθηκε. Τώρα η τροπολογία 122, άρχεται. Πέρας, απορρίπτεται 123 123 άρχεται πέρας απορρίφθηκε ισοψηφία πάλι απορρίφθηκε η 130 τροπολογία συγγνώμη η 125 η 125 τροπολογία άρχεται Πέρας. Απορρίφθηκε. Τοπολογία 130. Θα την ψηφίζαμε 126 Α, πρέπει να ψηφιστεί. Πρέπει να ψηφιστεί 126. Άρχεται λοιπόν. 126 είπαμε. Πέρας. Λοιπόν, για την 126 άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, για να το δούμε αυτό. Καταπίπτει. Ε, αν λέει 125 υιοθετηθεί. Δεν ψηφίστηκε. Γι' αυτό πρέπει να την ψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε την τροπολογία 126 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ναι κύριε Φερέρα, πείτε μας εσείς. Στον πίνακα ψηφοφορίας αναφέρεται ότι αυτή αποσύρθηκε. Όχι, στον πίνακα ψηφοφορίας δεν αναφέρεται ότι αποσύρθηκε. Θα ψηφιστεί σε περίπτωση που καταπίπτει η 125. Δεν αναφέρεται ότι αποσύρεται. Λάθος είναι σε σχέση με το Σταυρό. Σε αυτή την περίπτωση Ποια είναι η ένδειξη σε σχέση με τον εισηγητή. Εδώ είχαμε τον Σταυρό σε σχέση με αυτήν. Κύριε Φερέρε, άσχετα από τι ενδείξει ε, για την, για την ψηφοφορία, κάθε ένα έχει το δικαίωμα, κάθε ευρωβουλευτή να ψηφίζει όπω εκείνο κρίνει, άσχετα από τον πίνακα ψηφοφορία. Συγγνώμη κύριε Φερέρε, ακούστε με, η τροπολογία αυτή δεν αποσύρθηκε. Και όπω επιβεβαιώνει και η ίδια η κυρία Φράγκα που συνέταξε αυτήν, πρέπει να ψηφιστεί 126, γιατί 125 δεν εγκρίθηκε, έτσι, δεν εγκρίθηκε. Ναι κύριε Φερέρε, τι λέτε εσεί. Χωρί μικρόφωνο με μικρόφωνο σε αυτή την περίπτωση επειδή στον πίνακα ψηφοφορία είχαμε τον Σταυρό, μπορεί να υπήρξε, να παρισέφθησε κάποιο σφάλμα. Για κάποιου από του συναδέλφου είναι σημαντικό να ξέρουμε ποια είναι η σύσταση για την ψήφιση από πλευρά του Λέει η τροπολογία στο αρχικό. Απορρίπτει μια γενική μείωση του δυναμικού του στόλου με ε, συγκεκριμένο και δεσμευτικό τρόπο για κριτήρια, λόγω κριτηρίων της αγοράς η τροπολογία προτείνει να τροποποιηθεί η αρχική παράγραφος και η πρόταση της εισηγήτριας είναι να καταψηφιστεί αυτή η τροπολογία, έτσι, αυτή η πρόταση τροπολογίας. Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η τροπολογία όπως έχει συνταχθεί από την συντάκτρια. Περνάμε στην ψήφιση της τροπολογίας 126. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα, η τροπολογία 130 άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβαστική 19. Άρχεται. πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν εικοσιοκτώ. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 5 Ρέτζι. Ε, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 132 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 133 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 άρχεται. Πέρας.

Εγκρίνεται. 144 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 147 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 148 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 149. Άρχεται. Πέρασε εγκρίνεται 152 άρχεται 152 άρχεται πέρας απορρίπτεται 151 άρχεται πέρας απορρίπτεται 158 άρχεται πέρας εγκρίνεται συμβαστική 24 άρχεται πέρας εγκρίνεται εφόσον εγκρίθηκε 24 και η 158 η συμβαστική 24 δεν χρειάζεται να ψηφιστεί εφόσον είχε εγκριθεί 158. Οπότε θεωρείται ότι αυτή η ψηφοφορία για την συμβαστική 24 θεωρείται ως μη γενομένη. Οπότε πάμε στην προφορική τροπολογία που είναι συμβαστική με την 8 προφορική του κυρίου Γκάλαχερ για μια προσθήκη. Α, δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε.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 Πέρας. Απορρίπτεται. 156 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 157 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 159 Άρχεται πέρας. Απορρίπτεται. 160 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. Για την παράγραφο 8 η τροπολογία των ΦΑΜ ε, άρχεται. πέρασε. Εγκρίνεται. ΦΑΜ για την παράγραφο 9α καταπίπτει. Α. 161 άρχεται. 161 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 162 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 25 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 166 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 167 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 26 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 169 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 170 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 27 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Εκατόν εβδομήντα ένα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 177 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 28. Α, όχι. Α, αφού εγκρίθηκε 177, όχι. Yo creo que si las que decía que englobaba de las 100... Οπότε σα έλεγα 174 στην παράγραφο 17 καλύπτονται από τον 20, αλλά 28 δεν ψηφίστηκε. Γιατί είχε εγκριθεί 177. Οπότε δεν περιλαμβάνονται στην 28 αφού δεν υπάρχει. Άρα εγώ νομίζω ότι πρέπει να ψηφιστούν όλε οι παρακάτω. Vamos a ver. Que no, que. Τι όχι. Συμπεριλαμβάνονταν όλες σε μια συμβαστική που δεν ψηφίστηκε. Δεν καταλαβαίνω, λέει η κυρία Φράγα. Bueno, que están Πρόεδρος. Α, θεωρούμε ότι καλύπτονται λοιπόν. Α, ωραία, καλύπτονται. Καλύπτονται. Αφού μου λέει έτσι η γραμματεία, περνάμε στα 179. 179 άρχεται. Κύριε Φερέιρα. Ο κύριος... Κύριε Φερέιρα, παρακαλώ. κύριε Φράγα. Φράγκα. Έλα σπόδιν σε φτάδες. Ο κύριος Φερέιρα μπορούν να ψηφιστούν, δεν είναι ασύμβατες. Οι τροπολογίες που συμπεριλαμβανόντουσαν στο συμβιβασμό δεν είναι ασύμβατες με την 177, μπορούν να ψηφιστούν σε αυτό το βαθμό. Δεν είναι τεράστιο θέμα αυτό, δεν δίνω ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Φράγα. Κυρία Φράγα. Η 177 έχει αντικαταστήσει κάποιο τμήμα. Όλες οι άλλες τροπολογίες, κατά τη γνώμη μου λοιπόν, καταπίπτουν. Πρόεδρο, συμφωνείτε? Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Όχι, αλλά δέχομαι την απόφασή σας, εν πάση περιπτώσει. Αμίμε igual. Το ίδιο μου κάνει εμένα, λέει ο πρόεδρος. Δεν είναι καλά διατυπωμένος ο κατάλογος, γιατί αν συμπεριλαμβάνονταν στην συμβαστική που δεν ψηφίστηκε, τότε δεν συμπεριλαμβάνονται. 177 όμως αντικαθιστά την 28. Αλλά εάν δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όπως είπε ο εισηγητής, να περάσουμε στα 179. 179. Άρχεται. 179. Πέρας. Εγκρίνεται. 180. Πέρας. Εγκρίνεται. 181. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 182. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 183. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 184 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 29. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Άρχεται η Ρέτζι στη 12. Πέρασε. Εγκρίνεται. 189 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 194 άρχεται Πέρασε. εγκρίνεται οπότε τώρα περνάμε στη συμβαστική 30 τρία χωριστά τμήματα πρώτο τμήμα άρχεται 194 εγκρίθηκε. Α, οπότε όλα τα υπόλοιπα καταπίπτουν. Α, άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 31 τμήμα 1 άρχεται. Πέρασε εγκρίνεται. Συμβαστική 31 τμήμα δεύτερο, άρχεται, πέρας, εγκρίνεται. 201. Α, α, όχι, 198. 198, συγγνώμη. Πέρας. Απορρίπτεται. 200 άρχεται. Απορρίπτεται. 201 άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 202 άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 203. Άρχεται. πέρα. Εγκρίνεται. 204. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. ΦΑΜ στην παράγραφο 2 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 215. Α, συγγνώμη, 212. 212. 212. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 213. 213. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 33. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Ένα. Τροπολογία ένα. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δύο. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. τρία, Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. τέσσερα, Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. πέντε, Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική ένα, Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Έντεκα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δώδεκα άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεκατρία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 16 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 18. Πέρας. Εγκρίνεται. 19. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 24. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 25. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 26. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τριάντα. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 άρχεται πέρας εγκρίνεται 33 άρχεται πέρας απορρίπτεται 34 άρχεται πέρας απορρίπτεται συμβαστική 5 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. 40, συγγνώμη, 39, 39. Είναι συμβατή. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 38 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 41 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται 42 άρχεται πέρα. εγκρίνεται συμβαστική 6 άρχεται πέρας εγκρίνεται συμβαστική 7 άρχεται πέρας εγκρίνεται 45. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 48. Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 49. Άρχεται. Πέρασε. Απορρίπτεται. 50. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 51. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 52. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 53. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 54. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 55. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα το ψήφισμα όπως τροπολογήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφι υπέρ, 0 κατά, 3 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Φερέιρα. Περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία. Είναι η έκθεση για το πρόγραμμα πλαίσιο για την καινοτομία 2014-2020 ορίζον 2020 του κυρίου Τσουκαλά. Ξεκινάμε αμέσως λοιπόν, έτσι. Ωραία. Συνεχίζουμε. Τροπολογία 2. Έχετε όλοι έτσι τις τροπολογίες, τον πίνακα. Ξεκινάμε λοιπόν. Εντάξει, τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 21. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τοπολογία 22. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 27. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 28. Άρχεται. Πέρας απορρίφθηκε. Τροπολογία 32. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 34. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 35. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 37. Άρχεται. Πέρας απορρίφθηκε 38 άρχεται πέρας απορρίφθηκε τροπολογία συμβιβασμός 1 άρχεται πέρας εγκρίθηκε τροπολογία 42 άρχεται πέρας απορρίφθηκε τροπολογία 43 άρχεται πέρας απορρίφθηκε. Τροπολογία 49. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. 51. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Συμβιβασμός 2. Άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε. Τροπολογία 54. 54. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 55. Τροπολογία 55. 55. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία. Είναι γλωσσικό θέμα αυτό. Η 6 τώρα. Η 6, Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Συμβασμός 3. Άρχεται. Συμβιβασμός 3. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 8. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε τροπολογία 59. Συγγνώμη, δεν θα ψηφιστεί. 58. 58. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η 60. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 9 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. Η 10 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. Η 61 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. Η 62 άρχεται πέρας απορρίφθηκε. Η 11 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. Η 13 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. Η 63. Όχι, δεν θα ψηφιστεί. Ο συμβιβασμό 4 άρχεται πέρας. Εγκρίνεται. Η 65 άρχεται Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 13 άρχεται. Η 13 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η τροπολογία 67 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 14 άρχεται. Πέρας. εγκρίθηκε. Η 15 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Η 16 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Η 17 πέρας, εγκρίθηκε. Η 68 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Η 70 άρχεται, πέρας, απορρίφθηκε. Η 71 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Η 72 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Η 73 άρχεται, πέρας, εγκρίθηκε. Η 74 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. Η 19 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. Η 75 άρχεται πέρας. Εγκρίθηκε. 20 άρχεται πέρας εγκρίθηκε. Σκεπτικό, αιτιολογική σκέψη 1, τοπολογια 1 άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ψηφίζουμε την έκθεση, ε, την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε 21 ψήφοι υπέρ, καμία εναντίον, τρεις αποχές. Συγχαρητήρια. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο των ψηφοφοριών της ψήφισης για σήμερα το πρωί που είναι η έκθεση της κυρίας Πατράου για τα πτερίγια καρχαριών. Ξεκινάμε λοιπόν, εντάξει. Ξεκινάμε με την τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται τώρα. Τροπολογία 11. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε καταπίπτουν η NV9, NV8, η τροπολογία 20, η τροπολογία 22 τώρα άρχεται. Άρχεται. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε 22. Τροπολογία 13 καταπίπτει. Η τροπολογία 23, συγγνώμη, εσείς κυρία Πατράου, παρακαλώ. Πείτε μου παρακαλώ τι θέλετε. Sí. Ναι, παρακαλώ κυρία Πατράου, πείτε μας. Τίποτα, εντάξει, ωραία, ευχαριστώ. Τροπολογία 23 λοιπόν. Δεν θα την ψηφίσουμε γιατί απορρίφθηκε 22. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία επί της 14. Πέρας. Απορρίφθηκε. Η τροπολογία 15 άρχεται. Όχι, όχι, αφού απορρίφθηκε 14, όχι 15. Η ένβη 10. Η NV10 τώρα παρακαλώ. Άρχεται. NV10. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 24. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 25. Άρχεται. πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 27. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ένβι 12. Άρχεται. Πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 26 και τροπολογία 13 ένβη είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία επ' αυτών. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. Αιτιολογική σκέψη 2. Τροπολογία 1. Άρχεται. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Καταπίπτει NV11, τροπολογία 16. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. NV2, τροπολογία. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Τροπολογία 2. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 17. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 3. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 18. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 4. Άρχεται. Πέρας. απορρίφθηκε. Τροπολογία 19. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. NV4. Τρία λέει ο πρόεδρος. Συγγνώμη. NV4 βέβαια. NV4. Άρχεται. Πέρας απορρίφθηκε. NV5 άρχεται πέρας εγκρίθηκε. Τροπολογία 5 τώρα άρχεται. Τροπολογία 5. Πέρας τώρα. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 6. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 20. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία ένβη 6. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίθηκε. Ένβη 7. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 7. Άρχεται η 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 21. Όχι 21. Έτσι. NV8. Ποια έχουμε. Ούτε και η NV8. Έτσι. Δεν υπάρχουν άλλες τροπολογίες πια. Έτσι. Η τροπολογία 8. Ωραία. Η τροπολογία 8 λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 8. Ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Ναι. Πείτε μου, κυρία Πατράου. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Πατράου. Τροπολογία 8, λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 8. Ψηφίσαμε την τροπολογία 8 όπου είχαμε 15 υπέρ 8 εναντίον. Υπήρξε παρανόηση για το τι ψηφίζαμε. Παρακαλώ να επαναλάβουμε την ψηφοφορία, λέει ο κύριος Αρσένης. Μάλιστα. Νομίζαμε ότι ψηφίζατε την ένβη 8, λέει ο μιλητής. Λοιπόν, με κανένα τρόπο δεν ψηφίσαμε την NV8. Είπα τροπολογία 8. Η NV8 όπως αναφέρεται έχει καταπέσει γιατί εγκρίθηκε η 12, η τροπολογία 12. Έτσι λοιπόν δεν ψηφίστηκε η NV8, ψηφίσαμε την τροπολογία 8 με 15 υπέρ 8 κατά. Υπήρξε όμως παρανόηση λέγει ο κύριος Αρσένης να την ξαναψηφίσουμε. Πρόεδρο, εντάξει, ας επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Υπήρξε κάποι, από κάποιου ευρωβουλευτές κάποια παρανόηση, όχι από όλους. Το είπα με σαφήνεια εγώ, ψηφίζουμε την τροπολογία 8, όχι την ένδυ 8, τροπολογία 8. Τώρα λοιπόν ξαναψηφίζουμε, τροπολογία 8, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας. Τώρα καταψηφίστηκε. Τροπολογία 9 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 10. Άρχεται. Πέρας. Απορρίφθηκε. Με το ίδιο αποτέλεσμα. Ισοψηφία. Απορρίφθηκε. Μάλιστα. Κυρία Πατράου. Θα ήθελα να ζητήσω τα πρακτικά της συνεδρίας σας, της συνεδρίασης για την ε, τελική απόφαση για την ψήφιση. Γίνεται αυτό. Με αυτό το ίδιο αίτημα διατύπωσαν στην αρχή από άλλη ομάδα. Μετά κατανόησα από τις δικές σας ε, παρεμβάσεις τι επιθυμούσατε. Αν λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες, ε. δεν έχω κανένα πρόβλημα να δώσω τρία λεπτά να, να, να ξεκουραστείτε για να διαπραγματευτείτε και να επανέλθουμε. Εντάξει, σε τρία λεπτά. Συνεχίζουμε, αν συμφωνείτε λοιπόν, παρακαλώ, τη συνεδρία. Si les Αν συμφωνείτε μετά από αυτό το διάλειμμα να συνεχίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα την πρόταση. Ναι κύριε Ασένη, τι θέλετε να πείτε. Λοιπόν, έχουμε νομοθετικό θέμα, τεράστια παρανόηση για αυτή την νομοθεσία. Διαγράψαμε την εξαίρεση. Κάνουμε λόγο όμως για εξαίρεση στο κείμενο, εξαίρεση που δεν υφίσταται πια. Υπάρχει πλήρης ασυνέπεια και ασυμβατότητα εδώ. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία διαμαρτυρίες από τους άλλους. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε τη διαγραφή της εξαίρεσης. Ταυτόχρονα όμως από την άλλη πλευρά έχουμε αναφορά για μια εξαίρεση που δεν υφίσταται πλέον, μια και έχει διαγραφεί. Κύριε Αρσένη, μακάρι αυτό να ήταν η μόνη ασυμβατότητα που ψηφίζουμε σε αυτή την Επιτροπή εξάπαντος. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είδα εγώ αυτό και δεν το γνωρίζω. Δεν θα κάνουμε καμιά επανάληψη ψήφιση ε, ψηφοφορία όπω είναι λογικό. Θα συνεχίσουμε. Και αν στη συνέχεια από την, νομική υπηρεσία ή από τη γραμματεία ανακαλυφθεί ότι υπάρχει κάτι το μη συμβατό, ε, τότε θα το διευθετήσουμε. Είμαι πεισμένο ότι τα κείμενα που ψηφίσαμε για τι τροπολογίε ε, υπάρχουν πάνω από μία ή δύο, πολύ περισσότερε σε σχέση με μη συμβατά θέματα και απόλυτα αντιφατικέ τροπολογίε σε σχέση με το τι λέει η μία και η άλλη. Λοιπόν, πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια δουλειά σε ένα συνεκτικό κείμενο, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση λοιπόν όπως τροπολογήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίσατε όλες και όλοι πέρας ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα 11 υπέρ, 10 εναντίον, 3 αποχής εγκρίθηκε λοιπόν το ψήφισμα. Τώρα θα ψηφίσουμε την νομοθετική πρόταση στο σύνολό της. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας τώρα. Αποτέλεσμα εγκρίθηκε 12 υπέρ 9 εναντίον, δύο αποχές. Εγκρίθηκε λοιπόν η νομοθετική πρόταση. Συγχαρητήρια κυρία Πατράου. Περνάμε Λοιπόν, πέρα από την ευθυμία και τις χαρές που εκφράζονται, θα συνεχίσουμε γιατί καθυστερήσαμε πολύ. Έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Τώρα ως επόμενο σημείο και κλεισμένων των θυρών, παρακαλώ να φύγετε να αποχωρήσετε το δυνατόν ε, ταχύτερα εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται.